Meine Damen Κυρίες και κύριοι, σα σας καλωσορίζω θερμότατα σε αυτή την καταπληκτική αίθουσα που διαθέτουμε. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασής μας. Σχέδιο ημερήσια διάταξη, Ζητεί κανεί το λόγο. Όχι, ούτε αποφασίζει τη ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Προέδρου ακολουθούν. μου είπαν να σας αναφέρω και πάλι για το άρθρο 205 του κανονισμού μας. Το άρθρο 205 όπου ορίζεται ο ρόλος του διευρυμένου προεδρίου Δεν βλέπω τίποτα καινούριο, γιατί τι διαφορά έχει από αυτά που πάγια ακολουθούσαμε. Λοιπόν, προτείνω να συμφωνήσετε ότι ε, σας ενημέρωσα, λάβατε γνώση και μετά θα πάτε να το διαβάσετε και προσεκτικά. Ωραία. Πέτυχε και αυτό. Πάμε στο σημείο 3 τώρα. Παρουσίαση της εφαρμογής e-meeting λέει εδώ. Ηλεκτρονική συνεδρίαση. Όπω πρότεινε ο συνάδελφος Φλέκενστάιν, μήπω να φύγουμε και από την αίθουσα και να πάμε σε κανένα γρασίδι εδώ στην πλατεία Λουξεμβούργου να συνεδριάσουμε. Θα παρακαλούσα τους αρμόδιους να μας ε, μοιήσουν σε αυτά τα μυστικά. Ε, τα ονόματά σας. Ε, δεν ξέρω ποιος θα αρχίσει πρώτος. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το e-meeting, την ηλεκτρονική συνεδρίαση εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Αποθέσεων, Όπως ίσως γνωρίζετε, τώρα έχει μια πολιτική το Κοινοβούλιο για να μπορέσει να μειώσει την εκτύπωση των γράφων για τις συνεδριάσεις, γιατί πάρα πολύ συχνά τυπώνουμε, αλλά πετάγονται στον κάλθο των χρήστων αμέσως μετά την ε, συνεδρίαση ή ένα τμήμα μόνο αυτών χρησιμοποιείται, οπότε έχουμε πάρα πολύ διασπάθηση. Και αυτό αφορά λοιπόν και την ε, διανομή αυτών των εγγράφων. Πάντως είναι πολύ σημαντικά τα έγγραφα, είναι πάρα πολύ ζωτικό ε, τμήμα της, του κοινοβουλευτικού έργου, οπότε θα πρέπει να μπορεί και να τα βρει για να είναι προσβάσιμος και πιο νωρίς. Και βλέπετε τώρα εδώ Όσοι υποστηρίζει το Κοινοβούλιο αυτή την ε, εξέλιξη με αυτό το εργαλείο που λέγεται e-meeting ηλεκτρονική συνεδρίαση και αυτό τώρα και σας παρουσιάζω δύο λόγια. Πρώτα πρώτα για το, το περί τίνος πρόκειται, έχει σχέση με το ίντερνετ, εκεί βασίζεται, το αναπτύξαμε εδώ στο Κοινοβούλιο για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τις δικές σας και με εύκολο τρόπο μπορείτε έτσι να δείτε ηλεκτρονικά τα έγγραφα και αυτό μπορείτε να το κάνετε παντού, ανά πάσα στιγμή και με οποιαδήποτε ε, συσκευή. Θα πρέπει βέβαια να ξέρετε δύο-τρία πραγματάκια πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο εάν έχετε ε, μια κινητή συσκευή ε, θα ήταν πάρα πολύ σωστό τώρα να ε, την ανοίξει αυτή τη σχεδία και να ακολουθήσετε αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε. Επίσης, σας έχουμε μοιράσει ένα φύλλο, μια σελίδα που λέγεται Quick Start, εύκολος οδηγός δηλαδή για το e-meeting και εδώ μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του ε, διαδικτύου για να πάτε σε αυτό το σε αυτή τη σελίδα, σε, αυτή τη φάση το Quick Start και εκεί θα κάνετε login με ε, τους συνήθεις κωδικούς που χρησιμοποιείτε στο γραφείο σας ε, για τον υπολογιστή σας. Τώρα, με την άδεια του Προέδρου, θα πεθώ τώρα στον ε, συνάδελφο για να συνεχίσει την παρουσίαση αυτού του εργαλείου για τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Καλησπέρα, λέει ο άλλος κύριος. Ακριβώς όπως προαναφέρθηκε, αυτή η εφαρμογή ε, δεν χρειάζεται κάποιο είδους λογισμικό, απλώς χρειάζεται να έχετε σύνδεση ίντερνετ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ λοιπόν φτιάξαμε αυτό το shortcut, αυτό το, το σύντομο τρόπο πρόσβασης. Έχετε εδώ πέρα λοιπόν την επίσημη διεύθυνση του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, παρακολουθήστε, κάντε ό,τι κάνω. Λοιπόν, η διεύθυνση του Κοινοβουλίου, μετά κάθετος και μετά e-meeting σε μία λέξη χωρίς ε, διάστημα η τελεία και ε, τώρα βλέπετε ποια είναι η πύλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης. Βάζω εδώ τώρα τα δικά μου, λέει ο κύριος Φάντη, και βάλτε κι εσείς το δικό σας στη συσκευή σας. Αυτό λειτουργεί με το ασύρματο ίντερνετ, το Wi-Fi. Πάμε τώρα στο επόμενο. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα τις οδηγίες χρήσης. Βλέπετε αυτή την προσαγωγική σελίδα. Και εδώ αναφέρω ότι έχετε τρία βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνετε. Θα σας πω, πρώτα πρώτα μπορεί να διαλέξετε γλώσσα, επιτροπή και φυσικά την συνεδρίαση, την ημερησία διάταξη κλπ. Είμαστε τώρα στον χώρο που αποκαλούμε η meeting, υπάρχει όλες τις επιτροπές, άρα αυτό θα ισχύει για όλες τις επιτροπές. Βλέπετε εδώ αριστερά πώς μπορείτε να διαλέξετε την γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται η σελίδα, το παράθυρο που ανοίγει. Μετά διαλέγουμε την Επιτροπή, διαλέγουμε βέβαια την ΑΦΕΤ, εξωτερικών υποθέσεων, το σύστημα αυτό επισημαίνει ακριβώ τι σχετικέ πληροφορίε, τα δεδομένα και βλέπετε την τελευταία εκδοχή όλων των μεταφρασμένων εγγράφων. Ε, αυτά βέβαια ακόμα σε κάποιες επιτροπές ε, εκτυπώνονται, κάποιε άλλες είπαν ότι θα το σταματήσουν, αλλά τέλος πάντων αυτά τα παλιά τα τυπώνουν και τώρα τα έχετε σε μια σελίδα του υπολογιστή σας. Βεβαίω μπορείτε να κοιτάξετε και έγγραφα παλαιότερων συνεδριάσεων. Μπορούμε να πάμε επίση και μπροστά στο μέλλον, εάν υπάρχει ημερήσια διάταξη και αυτά μπορείτε να τα, βρείτε, εάν υπάρχουν στο, κάποιος τα έχει ανεβάσει στο σύστημα, άρα δεν υπάρχει θέμα αναμονή Εδώ δεξιά τώρα βλέπετε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 1 η Σεπτεμβρίου. Και πάμε τώρα στην 22η Σεπτεμβρίου το σύστημα θα βγάλει ό,τι πληροφορίες έχει η σημερινή συνεδρίαση. There is a plus sign in front of every item. Έχει βλέπετε αυτό το συν και μπορείτε τώρα είτε να αλλάξετε γλώσσα ε, ή μπορείτε να ανοίξετε κατά κάποιο τρόπο αυτό το, τον τίτλο, να δείτε τα παραπάνω πληροφορίες, να δείτε πληροφορίες για τον εισηγητή, Ό,τι τέλο πάντων πληροφορίε υπάρχουν σχετικέ με το έγγραφο αυτό. Και αυτό για όλες τις επιτροπές, για όλα τις συνεδριάσεις. Και τώρα ανοίγουμε το έγγραφο. μέσα σε διάταξη. Αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τη διαβάσουμε ή μπορούμε να ανοίξουμε τη σελίδα αυτή σε άλλη εφαρμογή. Εξαρτάται τι εφαρμογή έχετε εγκαταστήσει. Σαν χωρά κυκλοφορούν διάφορε εφαρμογέ, αυτέ διατίθενται, ούτω ώστε να είναι δυνατόν να διαβάσει κανεί το έγγραφο. Να είναι συμβατέ κατά με το έγγραφο. Ανοίγουμε τώρα λοιπόν, ανάλογα με το εργαλείο που θέλουμε. Εδώ λέει, ε, α, με αυτή την εφαρμογή μπορούμε να επισημειώσουμε κάποια πράγματα, ε, κάτι που είναι σημαντικό κλπ. Το έγγραφο αυτό που κατέβασα επιδέχεται σημειώσεις και οι σημειώσεις γίνονται, δηλαδή κατά επιτρόπο είναι το δικό σας αντίγραφο. Αυτά τα οποία κάνετε πάνω στο έγγραφο δεν μπορεί να τα δει ή δεν μπορεί να τα έχει κάποιος άλλος. Μετά βέβαια αφού τελειώσω την επεξεργασία ας πούμε του εγγράφου αυτού μπορεί κανείς να το διαβιβάσει ας πούμε στον συνεργάτη του με email σε κάποιο συνάδελφο και ε, επίσης όλες οι σημειώσεις που έχει κάνει κανείς ένα έγγραφο μπορεί και αυτές να τις ε, διαβιβάσει σε κάποιον άλλο. Α, βασικά αυτή είναι η πρώτη εκδοχή για το e-meeting και για αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε έγγραφο, να μπείτε μέσα στη σελίδα ας πούμε, να το σημειώσετε, να το αλλάξετε και να το δώσετε σε κάποιον άλλο και το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε επιτροπή. Να ας πούμε εδώ επιτροπή των προϋπολογισμών. Γιατί ακριβώ κάποιο βουλευτή μπορεί να δουλεύει σε δύο επιτροπέ και να χρειάζεται πρόσβαση σε δύο έγγραφα ταυτόχρονα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα του να βρούμε διάφορα σημεία της μέσης διάταξης τα οποία σχετικά με το σημείο της μέσης διάταξης μπορείτε να στείλετε ένα mail σε κάποιο συνάδελφο και γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν σύνδεσμο ακριβώς το σημείο της μέσης διάταξης που σας ενδιαφέρει. Αυτά για το e-meeting και το δύο για μια άλλη εφαρμογή που λέγεται e-committee, που είναι σχετική με το e-meeting. E-committee, ηλεκτρονική συνεδρίαση. Είναι κάπως πιο περίπλοκο σαν εφαρμογή. Εκεί περιέχονται όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με όλες τις επιτροπές. Βλέπετε το μενού πάνω-πάνω, βλέπετε τον σύνδεσμο προς το ε, e-committee. Οπότε πάμε στο AFET Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε όλες τις επιπλέον πληροφορίες. Και εδώ, όπως βλέπετε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίε πληροφορίες για σχέδια εκθέσεων των νομοδοτήσεων κλπ. Οπότε απλώς το να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή και είναι χρήσιμο εργαλείο να το ξέρετε. Να, ό,τι πληροφορίες έχουν να κάνουν με, το έργο κάποια επιτροπή. Αν κάποιο έχει ερώτηση, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εάν κάνουμε οικονομίες επειδή δεν τυπώνουν, θα μας φέρνουν ξανά καφέ αφού έχουμε εξοικονομήσει από εκεί χρήματα. Θέλει κανεί το λόγο. Ο Τσαρλ Ντάνοκ, παρακαλώ. Um, Στο τηλέφωνο Android δουλεύει. Γιατί έχω ένα Sony Xperia ε, που φτάνει μέχρι το επιλέξτε επιτροπή. Είναι έτσι πολύ σοφιστικέ. Από εκεί και κάτω φταίει το δικό μου τηλέφωνο, το Android της φταίει. The, is to work Υποτίθεται ότι λειτουργεί σε όλες τις ε, συσκευές, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να το δούμε και να το λύσουμε. Μια παρατήρηση μόνο. Είναι πολλά τα έγγραφα ε, που μπορούμε να βρούμε εκεί ε, και δεν χρειάζεται να τα έχουμε όλα εδώ τυπωμένα, αλλά πιστεύω ότι όταν έχουμε το τελικό σχέδιο της ε, έκθεσης και έχουμε και ψηφοφορίες για τροπολογίες, καλό είναι να τις έχουμε και γραπτός όταν ψηφίζουμε. Γιατί πολύ συχνά στις τροπολογίες και τέτοια πράγματα υπάρχουν συνάδελφοι που συναντούνται έξω στο διάδρομο με ένα στυλό, ένα μολύβι και προσπαθούν να κάνουν συσβιβαστικές. Και είναι και ένα θέμα πολύ πρακτικό επικοινωνίας αυτό και μέχρι τελευταία στιγμή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σε έγγραφη, σε έντυπη μορφή για να διαπραγματευόμαστε. Τώρα πρέπει να τρέχει ο καθένας με το iPad, με το iPhone, να κάνει μια διαπραγμάτευση στο διάδρομο. Φοβούμε ότι αυτό βλάπτει την επικοινωνία, επικοινωνία με την έννοια του μιλάμε και συζητάμε μεταξύ μας. Μόνο να τρέχουμε τις συσκευές δεξιά και αριστερά. Έχετε να πείτε τίποτα από αυτού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.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 Κοιτάξτε, το e-meeting είναι μία application, μία εφαρμογή την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Μπορείτε εσείς να αποφασίσετε σε επίπεδο δικής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τι είναι αυτό το οποίο θα δώσετε ε, σε ε, έγγραφο, σε χαρτί. Ε, υπάρχουν κάποια έγγραφα όμως τα οποία δεν είναι κατάλληλα όντως για smartphones και για τέτοιου είδους συστήματα συσκευές. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει ε, να ε, ε, δούμε κατά πόσον μπορούμε να συνδυάσουμε τη χρήση. Η απόφαση είναι δικιά σας, δηλαδή ποια έγγραφα θα είναι σε χαρτί, ποια θα είναι σε ταμπλέτες κτλ. Κύριε Τεχνική ερώτηση. Φαντάζομαι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι βαθμιαία να βγάλουμε το χαρτί ε, μέχρι πότε θα έχουμε ακόμα δυνατότητα χρήσης χαρτιού και δεν θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ε, την ε, ηλεκτρονική μορφή. Απάντηση. Η απόφαση είναι δικιά σας αφορά τη δική σας επιτροπή. Δεν υπάρχει ακόμα ε, συνολική απόφαση σε επίπεδο κοινοβουλίου ε, για να φύγει τελείω το χαρτί από χρήση, ε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλίου δεν υπάρχει τέτοιο είδου απόφαση. Εμεί προσφέρουμε αυτό το εργαλείο τώρα, αυτή τη δυνατότητα, αργότερα στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν και συσκευές για τα μέλη που θα στηρίζουν ε, εργασία η οποία θα χρησιμοποιεί όσο γίνεται λιγότερο χαρτί, αλλά επαναλαμβάνω ότι η απόφαση είναι δικιά σας, ανήκει στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή. Yes, in fact... Κοιτάξτε, ε, είναι ένα τεχνικό πρόβλημα ε, και βρήκαμε ε, τεχνική λύση. Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου και σημαίνει ότι λύνουμε σιγά σιγά τα προβλήματα. Το το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σιγά σιγά, να ακολουθήσουμε τα διάφορα βήματα ε, με απλό ρυθμό, όχι πολύ εντατικό. Γι' αυτό ακριβώς ε, κάνουμε και προτιθέμεθα να κάνουμε συνεδριάσεις ε, συμβουλευτικού έτσι, πληροφοριακού χαρακτήρα. Οποτεδήποτε θέλετε και εσείς μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθειά μας να σας κάνουμε μια τέτοια συνεδρία. Σε ευχαριστώ. Θα πρότεινα να το συζητήσουμε αυτό στο διευρυμένο Προεδρείο. Τι θα επιλέξουμε ως πρακτική για την ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπή και να ζητήσουμε από τη γραμματεία να ε, έχουμε και έγγραφα. Θα το συζητήσουμε, πάση περιπτώσει, και θα βρούμε κάποια λύση. Χρήσιμο είναι ως εργαλείο πάντως, διότι προφανώς δεν έχει νόημα να τυπώνουμε και τα πάντα. Εκεί θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό συμβιβασμό για να μπορούμε να λειτουργούμε και να εργαζόμαστε καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τη Γραμματεία να κάνει τις προτάσεις και να το συζητήσουμε στο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και περνάμε στο επόμενο θέμα, στη μέση διάταξη, υπαριθμών 4. και πέντε, νομίζω μαζί μπορεί να γίνει συζήτηση, έτσι δεν είναι. Μαζί και τα δύο θέματα. Σε αυτό το στάδιο της συζήτησης νομίζω είναι σκόπιμο να τα συζητήσουμε μαζί. Για τη Μολδαβία πρόκειται. Έχουμε αντίστοιχη κατάσταση με την Ουκρανία και εκεί. Διότι και εδώ πιέζει ο χρόνος. Βέβαια με την εξή διαφορά που είναι και αποφασιστική. Η Μολδαβία έχει ήδη κυρώσει τη Συμφωνία Σύνδεσης. Οπότε είμαστε τώρα στο στάδιο το επόμενο. Και το Νοέμβριο έχουν εκλογές. Οι Ρώσοι μέχρι και κόμματα ιδρύουν και τα χρηματοδοτούν. Και ασκούν και τεράστια πίεση. Και έχει νόημα πριν τις εκλογές θα πρέπει να ακυρώσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Σας έχω δίνει μία επιστολή που έλαβα σήμερα από τον Επίτροπο κύριο Φούλε και παρακαλεί και ο ίδιος ε, την έγκριση αυτή και την επικοινωνία. Θα παρακαλούσα να ακούσουμε τον εισηγητή να το φροντίσει. Πότε είναι εκλογές? Στις 30 Νοεμβρίου. Και θα πρέπει να το ψηφίσουμε στη μήνυ σύνοδο του Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, που είναι αρχές Νοεμβρίου. Έχουμε λίγο χρόνο. Και ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με την Ουκρανία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και εκεί να συντονιστούμε ε, χρονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό και μπορούμε να είμαστε και επικοδομητικοί. όπως έγινε και στην περίπτωση της Ουκρανίας που είχαν πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Αουστρεβίτσιους που είναι και εισηγητής για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά θα σας μιλήσω για, τις, ε, για το προσχέδιο συστάσεων όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου ε, σε σχέση με την Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με την της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μαλλοντομικής Ενέργειας ε, αφενός και τη Δημοκρατία της Μολδαβία ε, αφετέρου που ακολουθείται από μη νομοθετικού περιεχομένου ψήφισμα όσον αφορά τα την, ε, την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφενό και τη Δημοκρατία της Μολδαβία αφετέρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Μολδαβία είναι από πολύ μακρό χρόνο εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε μια λίγο διαφορετική κατάσταση και από γεωπολιτική και από οικονομική αλλά και από άλλες απόψεις. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι πάρα πολύ ε, απλός και απότομος. Εγώ προτείνω ε, την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας ε, από τη στιγμή που η Μολδαβία πρόκειται για έναν εταίρο στην ανατολική εταιρική σχέση, η οποία, ο εταίρο ο οποίος έχει δείξει ικανοποιητική στάση από πολλά χρόνια. Πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση στη Μολδαβία τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια χώρα ουραγός και τώρα είναι μια χώρα η οποία τα καταφέρνει πολύ καλά όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και επομένως πρέπει πραγματικά να την επενέσουμε για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, η γεωπολιτική κατάσταση είναι πλέον εντελώς διαφορετική από αυτήν που είχαμε παλαιότερα θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε και αυτή τη διάσταση υπόψη μας και να μην χάσουμε το χρόνο μας ε, με ε, πολλές και μακρές συζητήσεις. Με την ευκαιρία, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ε, να σας δώσω κάποιες αδρές γραμμές του, της έκθεσής μου ε, όσον αφορά αυτή τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ε, Βεβαίω ε, καλωσορίζουμε την υπογραφή αυτής τη συμφωνίας γιατί θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα στην διαδρομή που έχουν ήδη διανύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Μολδαβία και θα σημάνει βέβαια μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική και εμπορική συνεργασία. Υπογραμμίζουμε ότι η υπογραφή και κύρωση της συμφωνίας δεν αποτελεί βεβαίως τελικό στόχο περσέ, ωστόσο αποτελεί, ένα μέρος, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπό το άρθρο 49 η Μολδαβία όπως και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική και επομένως θα μπορούσε ε, να υποβάλει αίτηση ε, για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την προϋπόθεση ότι σέβεται τις θεμελιώδεις τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των μειονοτήτων κλπ. Στο προσχέδιο έκθεσης υπογραμμίζεται ότι εμείς θέλουμε αυτήν την συμφωνία για το καλό ολόκληρου του πληθυσμού της ε, ε, Μολδαβίας. Καλωσορίζουμε την, ε, το χρονοδιάγραμμα της σύνδεσης ε, που στόχο έχει τον υπερκερασμό των ε, προβλημάτων ε, και βεβαίως να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την περαιτέρω συνέχιση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Μολδαβίας πρέπει να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που επιτύχαμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό ακριβώς υπογραμμίζουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, ε, αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης η Μολδαβία όσον αφορά την χρηματοδότηση που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, καλούμε τα συμβαλόμενα μέρη να αναγνωρίσουν τις ανάγκες κατάρτισης οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν στην Μολδαβία. Μολδαβία, έτσι ώστε η Μολδαβία να γίνει ικανή να εκπληρώσει υποχρεώσει στο πλαίσιο τη συμφωνία και τη ατζέντα. Τονίζει επίση τη σημασία που έχουν οι ενίσχυση τη σταθερότητα, τη ανεξαρτησία και τη αποτελεσματικότητα των θεσμών, που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώ επίση και την εδραίωση του συστήματο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ευθεριών. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ιδιαίτερω να υπογραμμίσω ότι η Μολδαβία είναι, έχει πλέον διοικητική ικανότητα εντελώς διαφορετική από αυτήν που είδαμε ε, πριν από μερικά χρόνια και που την οδήγησε σε αυτή τη φάση σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις μολδαβικές αρχές να ε, ε, προετοιμάσουν τις επερχόμενες εκλογές ε, υπό το φως της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουν τα πολιτικά κόμματα και με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Επίσης υπογραμμίζουμε την ανάγκη, αναφέρω στο άρθρο 78, του, ε, την τροποποίηση του άρθρου 78 του Συντάγματος της Δημοκρατίας Μολδαβίας σχετικά με την εκλογή του Προέδρου, έτσι ώστε να μην ε, υπάρξει ξανά θεσμικό αδιέξοδο, το οποίο θα ήταν επιζήμιο για το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Και ζητεί να γίνει οποιαδήποτε σταματή μεταρρύθμιση σε συνένεση με την Επιτροπή της Βενετίας και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. Επίσης, ε, καλεί την ε, Μολδαβία να ενισχύσει την ε, αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ε, και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων δε και την πλήρη εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης που εντύχθηκε το 2013. Καλεί τις μοντανικές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι μηχανισμοί που ανήκουν στο σύστημα καταπολέμησης διαφθοράς, κυρίως δε το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης Διαφθοράς και το Εθνικό Κέντρο για την ακαιρεότητα, να χρηματοδοτούνται σωστά ε, και να έχουν το σωστό προσωπικό χωρίς αδικαιολόγητες επιρροές. Επίσης, καλεί τις μοδαβικές αρχές να διερευνήσουν σωστά και πλήρως όλες τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως δεν να αντιμετωπίσουν το θέμα της ατιμορρησίας σε περίπτωση κακομεταχείρισης και βασανισμών. Σημειώνουμε επίσης την σημασία της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων ε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα και η προστασία όλων των μειονοτήτων, κυρίως δεν αφορά τα άτομα ΛΟΑΔ. Επαναλαμβάνουμε επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί και να προωθηθεί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού, καθώς επίσης και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και, και η ουδετερότητα των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Υποστηρίζουμε πλήρως την εφαρμογή καθεστώτο απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για του μολδαβού πολίτε, υπενθυμίζοντα ότι η Μολδαβία ήταν η πρώτη χώρα εταίρο τη ε, ανατολική Ευρώπη και πέτυχε αυτό το, που πέτυχε το στόχο αυτό καλεί τις Μολδαβικές Αρχές να, να λάβουν υπόψη την εμπειρία που έχουν ε, αναλάβει μέχρι τώρα. Καμία άλλη χώρα στην γειτονική περιοχή δεν έχει επιτύχει τα όσα έχει επιτύχει η Μολδαβία όσον αφορά και το επίπεδο και την ποιότητα της εφαρμογής τους. Σημειώνει επίσης η έκθεση την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα των τελωνιακών και συνοριακών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη συνέχιση της οριοθέτησης των συνόρων με την Ουκρανία λέει, υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο της επαγγελματικοποίησης και αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. Πολλές, όπως και πολλές χώρες της γειτονιάς, οπωσδήποτε θα πρέπει η Μολδαβία να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον ε, και να, ε, ε, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο πλαίσιο μέτρων τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της μολδαβικής οικονομίας. Στηρίζουμε πλήρως τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της, του ρωσικού εμπάργου κατά των μολδαβικών προϊόντων, δίνοντας μεταξύ άλλων οικονομική στήριξη, καθώς επίσης μέσω επέκταση και εμβάθυνση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Καλούμε τις πρωτεύουσε Κισινάου αλλά και το Τυρασπόλ να συνεχίσουν να συμμετέχουν υποδομητικά στη συζήτηση ε, για αναζήτηση αποτελεσματικής λύσης στη διάνεξη της υπερνηστερίας και ε, επίσης να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού. Τονίζει τέλος ότι το λεγόμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο 5 συν 2 για τις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα δεν έχει εξασφαλίσει λύση και καλεί επομένως την ύπατη εκπρόσωπο καθώς επίσης και την, την ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να επιδιώξουν ενεργά τη βελτίωση της διαδικασίας ώστε να λυθεί η διένεξη χάρη σε ένα μεγαλύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας ως μέσο για την εφαρμογή της συμφωνίας καθώς επίσης και της ατζέντα σύνδεσης και καλεί την Κομισιόν να εντείνει την παροχή βοήθειας και πραγματογνωμοσύνης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο εσωτερικός έλεγχος και η λογοδοσία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η κυβέρνηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος ε, της ε, συνεδριάσεώς μας σήμερα ορθώς είπε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να εν το χρόνο, χωρίς να σπαταλάμε και να χάνουμε χρόνο, να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Καλό λοιπόν την Επιτροπή να μην χάσει άλλο χρόνο και να ολοκληρώσει επομένως τη διαδικασία τον μήνα Οκτώβριο με τρόπο ώστε να έχουμε δυνατότητα ε, να ακυρώσουμε την συμφωνία σύνδεσης με την Μολδαβία τον Νοέμβριο, μάλιστα αρχές Νοεμβρίου, έτσι ώστε ε, να έχουμε λίγο χρόνο πριν από, την, ε, από τις εκλογές της χώρας αυτής. Στο Κισινάου πιστεύουμε αγαπητοί συνάδελφοι ότι θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε δυνατό μέτρο την φιλοευρωπαϊκή συμμαχία έτσι ώστε όχι μονάχα απλώς να υλοποιηθεί η συμφωνία σύνδεσης, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην αναμόρφωση της χώρας εν ευθέτω χρόνο και με το σωστό τρόπο. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πρέντα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Στρεβίσιους, για ε, τα δύο ψηφίσματα αυτά και για τις ε, εξηγήσεις που μόλις μας έδωσε. Θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή και πιστεύω κι εγώ ότι πρέπει να συνάψουμε και να υπογράψουμε συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδαβία, η οποία την τελευταία πενταετία έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες, τεράστιες, για να φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Ελπίζω όμως η συμφωνία σύνδεσης να μην είναι του ίδιου τύπου με την Ουκρανία. Τι εννοώ, να μην έχουμε ανισορροπίες και ανισότητες σε αυτή τη σχέση και τη συμφωνία. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, αυτό τον καιρό η Ρωσία ασκεί πολύ μεγάλη πίεση και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν και πολιτικές παρενέργειες. Είναι μοναδική κατάσταση, ίσως και παγκοσμίως, ένα σοσιαλιστικό κόμμα να τοποθετείται αριστερότερα στο πολιτικό φάσμα από ένα κομμουνιστικό. Δεν το έχω ξαναζήσει εγώ σοσιαλιστές που να είναι πιο αριστεροί από τους κομμουνιστές. Πρωτοφανές φαινόμενο. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε λοιπόν για τον πρώην στρατηγικό μας εταίρο, τη Ρωσία, ότι ε, επεμβαίνει και σε ό,τι αφορά τις εκλογές και αυτές γίνονται σε μια πολύ περίεργη ατμόσφαιρα. Ε, αστερισμό για να το πω κάπως έτσι προσεκτικά. Υπάρχουν όμως ανισχυτικές οικονομικές εξελίξεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχει εμπάργο στις εξαγωγές ίνου από τη Μολθαβία. Και μάλιστα πριν επιβληθούν οι κυρώσεις ε, για τα τρόφιμα στις υπόλοιπες χώρες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε η Ρωσία να επιβάλλει ένα πολύ σκληρό εμπάργο στην Μολδαβία για ε, ε, αγροτικά προϊόντα και είναι τεράστιες οι ζημίες. Λύση δεν έχει βρεθεί, έχει μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ μεγάλες οι παρενέργειες και οι αρνητικές επιπτώσεις. Ε, και από το Σεπτέμβριο και μετά η Ρωσία αποφάσισε να ε, καταργήσει το ελεύθερο εμπόριο με τη δημοκρατία της Μολδαβίας, πράγμα που θα έχει επιπτώσεις και στην οικονομία ε, και πάλι. Τέλος, πρέπει να πω και να τονίσω ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία των εκλογών του Νοεμβρίου και πιστεύω ότι το κοινοβούλιο μας θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπροσωπείται επιτόπου. Και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Νομίζω πήγε αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και καλό θα ήταν εκτός από την αντιπροσωπεία του ΑΣΕ να υπάρξει και δική μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σεγητά και είμαι πεπισμένος ότι θα συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά. Θα κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις, ε, τροπολογίες, θα καταθέσω τις επόμενες υπέρες, ημέρες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συμφωνώ γενικά με τον εισηγητή, τα εξαιρετική έκθεση του και η παρουσίαση αυτής. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και πρώτα πρώτα όμως να συγχωρούμε τον εισηγητή για το αξιόλογο έργο του. Πάρα πολύ θετικά τα όσα παρατήρησε και επίσης θα πρέπει να χαιρετήσουμε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Μολδαβία τα τελευταία χρόνια σε αφορά τις μεταρρυθμίσεις και συμφωνούμε συγκεκριμένα με τον εισηγητή εκεί στο σημείο που ανέφερε τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συμφωνούμε με το περιεχόμενο της επιστολής την οποία σήμερα έλαβαμε από τον Επιτροπο κύριο Φίλε. Επίσης είμαι πεπισμένη ότι στενότερος δεσμός με τη χώρα αυτή, στενότεροι δεσμοί τέλος πάντων σημαίνει περισσότερη σταθερότητα. Και όπως ακριβώς ήταν πάρα πολύ θετικό το μέτρο το οποίο λήφθη για τα διαβατήρια των ε, Μολδαβών και έχω αναλάβει μια ε, σχετική έκθεση. Έχει ευρωπαϊκή προοπτική η χώρα. Έχει τη Συμφωνία Σύνδεσης η οποία αποτελεί ε, βήμα εξυγχρονισμού, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κληθούν να προχωρήσουν ταχαίως στην κύρωση της σχετικής συμφωνίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Ακριβώ όπω τα λέτε και κύριε Ζηγητά στην αρχή. Η προεκλογική εκστρατεία επισήμω ξεκίνησε. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με τα καλύτερα των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και βεβαίω να εμεί ω παρατηρητέ να είμαστε εκεί, να στείλουμε την αντιπροσωπεία ε, του Κοινοβουλίου από όλε τι πολιτικέ πτέρυγε. Μια τέτοια αποστολή παρατηρητών και θα πρέπει επίσης να απευθυνθούμε στις αρχές της χώρας να συνεργαστούν με τους διεθνείς φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, κύριε Σιγητά, πάρα πολύ θετική θεωρούμε την υπογραφή της συμφωνίας της ε, συμμετοχής της χώρας για το ορίζον 2020. Και αυτό πρόκειται να βοηθήσει για, τον, για την καινοτομία, για την ανταγωνιστικότητα, για την ε, απασχόληση στη χώρα και επίσης όσον όλη την υπερδυνιστερία. Όπως είπατε, πρέπει να βρεθεί κάποια αποτελεσματική λύση, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε η συνάντηση 5 5-2 της Βιέννης ε, σχετικής ομάδας την περσμένη εβδομάδα. Χρειάζεται μακρόπνοη λύση και γι' αυτό και παρακαλώ όλοι οι εταίροι να κληθούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να προστατευτεί η εδαφική κυριότητα της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νάρτ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Αστροβίτσιος, για την έκθεση. Είναι πλήρης και είναι πάρα πολύ προσεκτική, σόφρον, ρεαλιστική. Ε, Ιδίω εκεί στο σημείο 20 που αφορά τις ε, επιθυμητές σχέσεις μεταξύ αυτών ε, των, μεν και των δε, δηλαδή του Τυρασπόλ και του Κισινάου. Επίσης όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτού του είδους η μόνιμη ένταση. Δεν είναι εδώ μια οποιαδήποτε γειτονική σχέση, είναι γειτονική σχέση με κάποιον πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα πρέπει και η Ευρώπη να συνεχίσει την επαγρύπνηση γιατί υπάρχει τώρα το σοβαρό γεγονός του συνορωσικού άξονα. Και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγιναν κάποια παράλογα πράγματα γιατί είχαμε την Βλαχία και Μολδαβία. Αυτά συναποτελούσαν την ε, Ρωμανία και κατόπιν προσθέθηκε η Τρανσιλβανία. Πάντως τώρα μιλούμε για κάποια τρίτη χώρα. Χώρα που είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέδρος πριν είπε για ο συνάδελφος μάλλον ο εισηγητής είπε για αυτού του είδους τις θεσμικές ε, διαστάσεις του θέματος, αλλά τόνισε και την οικονομική κατάσταση της χώρας που είναι οριακή. Όταν ήταν Σοβιετική Ένωση, έκανε εξαγωγές ε, τρακτέρ και αγροτικών προϊόντων, όλα αυτά όμως τελειώσαν τώρα. Τώρα η χώρα ε, φτωχοί. Και επομένως τώρα βλέπει αλλού, βλέπει προς την Ευρώπη. Επομένως γι' αυτό και θα πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις και να καταλήξει αυτή η πορεία στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, όχι, σε δύο. Στο σημείο 13, σημείο 13, εδώ υπάρχει μια πάγια μνήα και σωστά κατά τη γνώμη μου όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΔ. δεν είναι μια ούτε μειονότητα. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Και έχουμε και τους γκαγκαούς που είναι και αυτή σημαντική μειονότητα. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για μειονότητε μόνο για εκείνε οι οποίε έχουν κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό ε, πολιτιστικό, όπω οι Τούρκοι, τουρκική δηλαδή μειονότητα, ε, ή του ΛΟΑΔ. Εδώ πέρα έχουμε και αυτή τη γαούζους και για αυτούς θα πρέπει να εγγραφεί κάτι στο κείμενο γιατί είναι πολύ περισσότεροι από τους ΛΟΑΔ. Φυσικά από πλευρά ανθρωπιστική είναι το ίδιο σημαντική μειότητα. Τώρα παρακάτω. Στο σημείο 16. Στο σημείο 16 γίνεται μια θέματο που θεσμικά, στεγματικά είναι σωστό, αλλά εδώ πέρα δεν συνάδει προ την κατάσταση. Λέμε για τα σύνορα τα Μολδαβο-Ουκρανικά. Εκεί δεν έχουμε τόσο καλούς ελέγχους. Γιατί είναι κοινό το σύνορο με την υπερτινιστέρια, οπότε και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορεί να ελέγξει η Μολδαβία για το τι γίνεται σε αυτά τα σύνορα. Κάτι άλλο τώρα που θα θεωρώ σημαντικό. Για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις. Έγινε ένα βήμα πρόοδο πάρα πολύ σημαντικό. Όμως εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο πολύ πραγματικό. Αφορά κάτι το οποίο συμβαίνει. Πολλές φορές έχουμε εδώ διαπράξει εγκλήματο. Πολλέ φορέ έχουμε κάποιου που παίρνουν διαβατήρια και τα χρησιμοποιούν για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα. Η υπερδυνιστερία, όπω είναι λογικό, αναγνωρίζεται ως τμήμα της Μολδαβίας. Οποιοςδήποτε πολίτης ε, της υπερδυνστερίας μπορεί να ζητήσει και να λάβει όπως είναι λογικό το μολδαβικό διαβατήριο. Με αυτό το διαβατήριο, λόγω των ιστορικών ε, πασιών σχέσεων μεταξύ Μολδαβίας και Ρουμανίας, που δηλαδή μέχρι το 1945 αποτελούσαν ένα και μόνο κράτος, μπορούν να ζητήσουν για να λάβουν το ρουμανικό διαβατήριο. Άρα διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε το πρόβλημα το οποίο αναδύεται. Οποιοδήποτε από οπουδήποτε, εάν πάει στην υπερτινιστερία, μπορεί να αποκτήσει διαβατήριο της υπερτινιστερίας και μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω ρουμανικού διαβατηρίου, να αποκτήσει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σωστός έλεγχος ε, για το τι είδους θεωρίες δίνονται από και προς το ε, Κισινιόφ για να δούμε τι γίνεται με αυτούς ε, οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκλήματα μέσω της υπερδινιστερίας παίρνουν το μολδαβικό διαβατήριο και μέσω αυτού το ρουμάνικο και σε σχέση με αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και θα πρέπει επίσης να επαγρυπνούμε πάρα πολύ γιατί τώρα μιλούμε για μια, μια, μια περιοχή, μια χώρα, μια περιφέρεια που τα σύνορά της είναι διάτριτα. Ο πρόεδρος. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ναι. Είναι περίπλοκη εδώ διαδικασία και δεν συζητούμε για πρώτη φορά τις εξελίξεις ε, ούτε τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας δεδομένων και των εξελίξεων της τελευταίας διετίας, νομίζω, το θέμα της Συμφωνίας Σύνδεσης και ε, της ελευθέρων συναλλαγών αποκτά έτη ε, μεγαλύτερη σημασία. Ευχαριστώ πολύ για τα διάφορα σημεία που αναφέρθηκαν στο ε, ψήφισμα και τα ανέγνωσε ο εισηγητής. Θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που έχει να κάνει και με τη μελλοντική μας εργασία, θα μας απασχολήσει και αργότερα, δηλαδή στα πλαίσια της γεωργίας και το είχαμε συζητήσει και για την Ουκρανία. Στο σημείο 2 λέει ότι η υπογραφή και επικύρωση της συμφωνίας δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διαργασίας. Και στο 3 το συγκεκριμενοποιεί και λέει ότι βεβαίως και η δημοκρατία της Μολδαβίας δίνεται κάποια στιγμή να εγγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, το καλωσορίζω κάθε χώρα, ε, εάν το επιθυμεί η πλειοψηφία του πληθυσμού, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην Ένωση. Ε, βεβαίως, ε, με έλεγχο πάντα αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Πλην όμως, αυτή η διαδικασία επικύρωσης θα έρθει πριν τις εκλογές. Δηλαδή, με αυτή τη δήλωση εμείς αναμειγνιόμαστε σε μια άμυλα, σε έναν ανταγωνισμό που γίνεται εντός της χώρας για τις εκλογές. Διότι ο πληθυσμός, ο λαός αναμένει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία προθυμία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεύρυνση. Λοιπόν, είναι το, πώς να το πω, με τα λόγια είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι, αλλά στην πράξη μάλλον διστακτικοί. Η κυρία Χάνς και ο κύριος Βόλσκι, Σάριος Βόλσκι στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, είπανε «Βεβαίως θέλουμε η Ουκρανία να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πλειοψηφία λέγει ρητά όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, λοιπόν και έντιμοι. Άρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να παραμείνει, αν μπορεί να παραμείνει έτσι αυτή η διατύπωση, γιατί υπάρχουν και αγωνίες και προβληματισμοί και ανησυχίες και στα 28 κρατημέλη για μια νέα διεύρυνση ευρύτερη. Θα πρέπει να τα λέμε και εμείς ε, αυτά και με τρόπο πιο διαφανή και πιο ειλικρινά τα συζητούμε. Ένα επόμενο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το εξή. Με τη συμφωνία σύνδεσης και ακόμα περισσότερο της ε, ε, ελευθέρων και την Τετάρτη ε, θα το συζητήσει η Επιτροπή Ίντα, Διεθνούς Εμπορίου αυτό το θέμα, εκεί γίνεται σαφές ότι μιλούμε για την πραγματική ζωή των ανθρώπων, για την καθημερινότητα και την οικονομική τους κατάσταση που έχουν κατά μέσο όρο ε, μηνιαίο εισόδημα 100 ευρώ. Είναι πάρα πολύ φτωχή η χώρα, η φτωχότερη της Ευρώπης, με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν για μια τέτοια χώρα, μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών όπου η μολδαβική οικονομία εκτίθεται στον ανταγωνισμό απροστάτευτη ποια θα είναι η κοινωνική ε, κατάσταση, γιατί είναι και περιορισμένες οι εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας από άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ε, με την ε, κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών είχαν στο παρελθόν. Λοιπόν, τι γίνεται με τα τελωνία απέναντι στην Τελωνιακή Ένωση, που σημαίνει αύξηση των δασμών, οπωσδήποτε. Σε περίπτωση που η Μολδαβία είναι σε θέση και επιτρέπεται να εξάγει εμπορεύματα ε, στη Ρωσική Ομοσπονδία και στα άλλα κράτη που έχουν τελωνιακή ένωση. Ενώ η δική μας συμφωνία σημαίνει μείωση των δασμών. Αυτά λοιπόν τα θέματα που τα βρήκαμε μπροστά μας στην Ουκρανία τα ξανασυζητάμε για τη Μολδαβία και αύριο θα έρθουμε να τα ξανασυζητήσουμε για την Ουκρανία. Γεωργία, συγγνώμη. Λοιπόν, χρειάζονται μεταβατικές ρυθμίσει. Τι δυνατότητες μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα για να μην έχουμε μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και δεινά. Και ένα τελευταίο, βεβαίως είναι σημαντικό το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίων, αλλά και η υπερδνηστερία την Άνοιξη κατέθεσε αίτηση για ειδικέ σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ναι, είναι τμήμα της Μολδαβίας η υπερνηστερία, αλλά ξέρουμε και το ιστορικό προστσές και τη διαδικασία. Παλαιότερα ήταν Ουκρανία, μετά ενώθηκε με τη Μολδαβία. Ε, δηλαδή, ε, ε, Ρουμανία, Ουκρανία. Εδώ βγαίνει ο πρόεδρος της Ρουμανίας και λέει «Μα η Μολδαβία ουσιαστικά Ρουμανία είναι». Και πάλι μπαίνουμε σε αντιφάσεις και σε προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική στάση θα πρέπει να το σκεφτούμε και πολύ προσεκτικά να διατυπώσουμε ε, αυτή την έκθεση για να ε, αποφανθεί και το Κοινοβούλιο για αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του και εγώ πιστεύω ότι είναι μια έκθεση πολύ καλή και ε, στραμμένη προς το μέλλον. Πραγματικά νομίζω ότι εάν βεβαίως βρεθεί η πλειοψηφία ε, στο σώμα για τη Συμφωνία Σύνδεσης, αυτή να εκφραστεί ε, σαφώς πριν από τις ε, ευρωπαϊκές, συγγνώμη, μολδαβικές εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι Μολδαβοί να, κάνουν, ε, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να εκφραστούν από αυτή. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες στην έκθεση, οι οποίες αφορούν πάντως την ίδια γραμμή με αυτήν της αρχικής εκθέσεως. Να σημειώσω τα εξή όμως θα θέλαμε να υπάρχει μια παράγραφος η οποία να αναφέρεται την, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μερικής ενημέρωσης ε, που ε, ε, παρουσιάζουν έλλειψη πολυφωνίας και υπερβολική συγκέντρωση στα χέρια ενός ιδιοκτήτου. Θα θέλαμε επίσης να γίνει κάποια αναφορά στην ενεργειακή στρατηγική και θα θέλαμε να πούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το ε, Εθνικό Σχέδιο Δράσης 13-15 όσον αφορά την ενέργεια. Επίσης θα θέλαμε και μια γενικότερη αναφορά, ε, γιατί βεβαίως δεν είναι και η πρώτη φορά που θα, τελευταία φορά που θα γίνει ε, λόγος σε αυτά τα πράγματα. Πρώτον, λέω, να επενέσουμε το Κισινάου Απ' την άλλη πλευρά να πούμε ότι το πρόγραμμα ε, της ε, ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης έφτασε πλέον στα όρια του και επομένως θα πρέπει να μελετήσουμε και εδώ και γενικότερα στο σώμα κάποια νέα πρότυπα, κάποιες νέες αρχές όσον αφορά την Ανατολή, τις ανατολικές χώρες και την εταιρική σχέση και την πολιτική ανατολικής γειτονίας. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ εγώ και θα ήθελα καταρχάς να ε, ευχαριστήσω τον συνάδελφο ε, και να πω ευθύς εξ αρχής ότι συμφωνούμε ως ΕΛΚ με τη σύσταση του να ακυρώσουμε τη συμφωνία. Νομίζω ότι αυτόν τον καιρό και λόγω της ρωσικής πίεσης στα γειτονικά κράτη είναι το σωστό μήνυμα αυτό για μας. Για να σταλεί και προς την κατεύθυνση της Μόσχας. Σε σχέση με αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην έκθεση. Θα αναφερθώ σε συντομία γιατί κάποιος συνάδελφος αναφέρθηκε στους γκαγκαούζους. Όντως, αν ασχοληθεί κανείς εκτενέστερα. Φαίνεται ότι η Μολδαβία είναι μικρογραφία Σοβιετικής Ένωσης κάπως. Υπάρχει και μια ιδιάζουσα πραγματικότητα που έχει αναπτυχθεί εκεί. Και επειδή ενδεχομένω μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, το οποίο και έξωθεν να οξυνθεί, καλό θα ήταν να πούμε κάτι κι εμείς. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να μιλάμε για κόπωση διεύρυνσης γενικά, enlargement fatigue, ε, και να μην αναφέρουμε το άρθρο 49, διότι υπάρχουν και κάποιοι χρονικοί ορίζοντες που είναι τόσο μακρινοί, ώστε να μην καλύπτονται με κάποια επίκαιρα επιχειρήματα. Δεν λέμε δηλαδή να μπει η Μολδαβία στην Ένωση μέσα στα επόμενα πέντε έτη. Είναι άλλοι χρονικοί ορίζοντες εδώ και οι περίοδοι για τις οποίες μιλούμε. Και θα ήταν λάθος μήνυμα να μην αναφέρουμε το άρθρο 49 και προς τη Μόσχα και πάλι, ότι έχουμε κουραστεί να διευρυνόμαστε. Βεβαίως έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι πολύ σκληρή αυτή η διαδικασία μετάβαση και μετασχηματισμού της χώρας, που έρχεται να επιδεινωθεί και από το μποϊκότ της Ρωσίας και για το εμπόριο και για τα εμπορεύματα. Έχει λοιπόν σημασία πολιτική να γίνουν σωστά οι μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου, οι διοικητικέ και γενικότερα των θεσμών. Και στο παρελθόν γνωρίσαμε θετικές εξελίξεις, οι οποίες κάπως ε, επιβραδύνθηκαν στη συνέχεια. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία τώρα να επιμείνουμε εμείς αυτό. Και ελπίζω να φτάσει το θέμα και γρήγορα στην Ολομέλεια πριν τις βουλευτικές τους εκλογές, δηλαδή τον Νοέμβριο, να έχουμε καταφέρει και προλάβει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα. Υπάρχει λόγος όμως να επαγρυπνούμε και χρειάζεται προσοχή, γιατί μένουν 69 μέρες ακόμα. Όταν... Αν σκεφτείτε πότε τέλειωσαν οι ελβιακοί αγώνες στο Σότσι και πότε έγινε η κατοχή στην Κρυμαία, ήταν λιγότερες από 50 μέρες, δηλαδή 69 μέρες είναι πολύς χρόνος. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει μια πρόοδος και επειδή αναφέρθηκε και κάποιος άλλος στο θέμα του πότε και ρωτάω και τη γραμματεία για τη γεωργία. Πότε επίκειτα η ίδια συζήτηση και ψηφοφορία. Ξέρουμε περίπου έτσι για να προσανατολιστούμε χρονικά. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή για το ισορροπημένο και ορθολογικό περιεχόμενο των δύο κειμένων του. Δράτομαι της ευκαιρίας για ε, να αναφερθώ θετικά στην επιστολή που εστάλει από την Επιτροπή μας στον, Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για τη διεύρυνση αυτού αυτό ε, το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία της δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μη λησμονούμε ότι έχουμε εκλογές στη χώρα αυτή στις 30 ε, Νοεμβρίου. Ως μέλος της αντιπροσωπείας για την ε, Μολδαβία θα ήθελα εδώ να αναφερθώ επενετικά στις μεγάλες προόδους που έκανε αυτή η μικρή χώρα τα πέντε τελευταία χρόνια ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πολλές προόδους κατάφερε να ε, επιτύχει η ε, Μολδαβία όπως ας πούμε απελευθέρωση και η απελευθέρωση ε, των θεωρήσεων ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό και ευχαριστώ εν παρόδο την κυρία Φαγιόν για την θετική προς την κατεύθυνση αυτή έκθεσή της. Όσον αφορά τώρα τις, ε, τις, ε, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, ε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτής της συμφωνίας για, τις, για τις πολιτικούς αυτούς σχηματισμούς και είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Πρέπει εμείς να καλέσουμε όμως όλες τις πολιτικές ομάδες, όλα τα πολιτικά κόμματα ε, να ε, δραστηριοποιηθούν σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Προλαλήσαντες ε, ομιλητές αναφέρθηκαν στον, στο θέμα το οποίο αφορά την απόκτηση ρουμανικής ηθαγένειας από τους πολίτες της, της Μολδαβίας. Πρέπει να σας πω ότι η απόκτηση της ηθαγένειας ε, αφορά μονάχα το γιου sanguinis», δηλαδή μονάχα αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι οι γονείς τους ε, ή οι παππούδες τους ε, είχαν ρουμανική υπηκότητα, τότε μόνο μπορούν να αποκτήσουν και εκείνη τη ρουμανική υπηκότητα. Επομένως θεωρώ ότι είναι υπερβολικές αυτές ε, οι αναφορές ε, στην εγκληματικότητα ε, της υπερνηστερίας και της, αυτού, του κινδύνου ας πούμε να περάσουν εγκληματίες στα σύνορα λόγω ακριβώς αυτών των διαβατηρίων. Θα ήθελα τώρα να πω και κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα Ακούσαμε τον επικεφαλής ε, των ε, στρατιωτικών δυνάμεων ε, της Ευρώπης ε, να λέει ότι αυτή, αυτός ο υβριδικός πόλεμος που είδαμε στην Ουκρανία ε, υπάρχει κίνδυνος να ε, προχωρήσει και στη Μολδαβία. Βεβαίως υπάρχει κάποιος κίνδυνος, βεβαίως υπάρχουν προκλήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παρόντες για να βοηθήσουν τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κύριε Σιγητά. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι η δεξιά όταν μιλάει για εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ Άκουσα ε, τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ να μιλάει για μικρογραφία της Σοβιετικής Ένωσης ή να ε, βιαστούμε μη τυχόν και κάνει τα ίδια με την Κρυμαία η Ρωσία. Λες και δεν έχει αυτό καμία σχέση με τις εθνικές μειονότητες ή τις μειονότητες ΛΟΑΔ. Έτσι καταλαβαίνόμαστε πολύ καλύτερα όταν συζητούμε και τη συμφωνία της Μολδαβίας και τι σημαίνει. Στη χώρα μου υπήρχε ένα group punk ε, όταν ήταν ο ψυχρός πόλεμος και είχε ένα τραγούδι με ένα τίτλο «Τι θα έκανες αν επιτεθόταν η Σοβιετική Ένωση» και αυτή η Επιτροπή κάθε φορά μου θυμίζει το Stanley Kubrick και την περίφημη ταινία ε, ε, ε, Dr. Strange που είχε ένα θάλαμο επιχειρήσεων και σχεδίαζε πώς θα επιχειρήσει και πώς θα επιτεθεί στη Ρωσία. Η κατάσταση λοιπόν στη Μολδαβία δεν είναι όμορφη, είναι από τις πιο φτωχές στην Ευρώπη από τις 187 στην ανθρώπινη ανάπτυξη είναι 111, 61 για τους άνδρες και 69 ε, το προσδόκιμο ζωής ε, για ε, τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες εξωθούνται στην πορνεία, στις σεξουαλικές αγορές στην Ευρώπη. Ένα από τα τρία παιδιά στη Μολδαβία εμφανίζουν εγκεφαλικές βλάβες λόγω έλλειψης ιωδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γιατί έχει γίνει για να βοηθήσει όλο αυτό τον κόσμο. Όχι. Ο κύριος Μακέιν είχε δίκιο όταν είπε πριν από λίγες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να ξαναμπούν τα συστήματα στη Τσεχική Δημοκρατία και στην Πολωνία ε, τα αντιπυραυλικά και η Μολδαβία και η Γεωργία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Γιατί μας έχει πιάσει αυτή η βιασύνη να κυρωθεί πριν μπορέσουν να ψηφίσουν οι Μολδαβοί. Το 2009 ε, ήταν σκεπτικιστές αυτοί που επικράτησαν απέναντι στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοψηφίσματα δείχνουν ότι οι πολιτικές δυνάμεις που είναι κατά της συμφωνίας ε, φιλίας ή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλειοψηφούν ενδεχομένω. Και ρωτώ τόσο πια ε, μας πείραζε τέτοιο πρόβλημα έχουμε να περάσουν εκλογές και μετά να κυρώσουμε. Γιατί αυτή η βία δεν έχω καταλάβει. Κύριος Φλέκενστάιν, τρία σύντομα. Πρώτον, η αναφορά στο άρθρο 49, νομίζω θα πρέπει να τη χειριστούμε εξίσου πραγματιστικά και ρελεστικά όπως έγινε και με την Ουκρανία. Είτε είτε. Δηλαδή δεν μπορούμε στο ένα ψήφισμα να το βάζουμε και στους άλλους όχι. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε πάντα, όταν το συζητάμε και με τους φίλους εκεί, ότι είναι μακροπρόθεσμη προοπτική, έτσι δεν μιλούμε για αύριο, το για μεθαύριο. Δεύτερον, προφανώς είμαι υπέρ της κύρωσης, απλώς θέλω να ρωτήσω πότε ε, προτίθεται να μας ενημερώσει ο κύριος Ντεχούχτ. Μήπως να το, θα το ξανασυζητήσουμε με τη Ρωσία, ε, μήπως να μην τον περιμένουμε τον κύριο Ντεχούχτ. Γιατί Γιατί για την Ουκρανία είναι σκόπιμο να συνεννοηθούμε με τη Ρωσία για τις πιθανές επιπτώσεις, ενώ για τη Μολδαβία όχι. Και ποια είναι η διαφορά. Θα με ενδιαφέρε, εμεί ζήσουμε και νέες εκπλήξεις. Τρίτον, δεν υπάρχει άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μιλεί για ένταξη της Μολδαβίας στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, ο Μακέιν είναι πουμπλικάνο, είναι και έχει και προεκλογική εκστρατεία, δεν χρειάζεται εμεί να τα υιοθετούμε αυτά, αυτά που λέει το Tea Party δεν τίθεται αυτό στην ημερήσια διάταξη, δεν είναι θέμα προσυζήτηση. Και ένα τελευταίο που δεν έχει καμία σχέση με την Επιτροπή μας εδώ, αλλά θα παρακαλούσα στο βαθμό που σας αφορά να με υποστηρίξετε. Την Πέμπτη, την πέμπτη η Euronest για πρώτη φορά θα συσταθεί αυτή η μεγάλη δική μας αντιπροσωπεία για την Ανατολική Γειτονία. Και θα σας παρακαλούσα να με βοηθήσετε όσο γίνεται να μην συνεδριάσουν όλες οι επιτροπές τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, ε, της Euronest εννοώ, αλλά τουλάχιστον μία στη Γεωργία και μία στη Μολδαβία. Έτσι ακριβώς για να δείξουμε ότι συνεργαζόμαστε, υπάρχει παρουσία, μπορεί να είναι και δημόσια, ε, εάν θέλετε, για να μην λέμε ότι είναι μόνο λόγια στα χαρτιά, αλλά ότι αποκτά σάρκα και ως τα αργά, αλλά σταθερά. Αυτά, ευχαριστώ για το τελευταίο παρακαλώ για την υποστήριξή σας. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχουν οι κανόνες ότι δεν ταξιδεύουν αυτές οι επιτροπές, ε, να το φροντίσουμε. Thank you, Mr. Chairman. I, really just... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κάρβερ. Θα σας πω ότι έχουν να ζητήματα Ναι, η σχέση με τη Ρουμανία είναι σημαντική που είναι και θα πρέπει και εμεί σοβαρά να προβληματιστούμε για το τι γίνεται όσον αφορά για τα μαντάτα για την διαφθορά στη Ρουμανία. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά τα διαβατήρια τα οποία πουλούνται σε κάποιου που μπαίνουν από την Μολδαβία. Και είπαμε ότι μπορούν να μπαίνουν Μολδαβοί και να αγοράζουν διαβατήρια από τη Ρουμανία λόγω των στενών σχέσεων των δύο χωρών. Και έτσι υπάρχει μια κερκόπορτα προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει τόσο ο πύρετο τη διεύρυνση. Το θέμα δεν είναι να αφήσουμε έξω την Μολδαβία. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με την Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Ο κόσμο λέει ε, ότι έχουμε τόσα προβλήματα με τη Ρωσία και άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί αυτά τα οποία κάνουμε εμείς δεν βοηθάνε την κατάσταση. Νομίζω ότι το timing που προσπαθούμε τώρα να εφαρμόσουμε για τη Μολδαβία είναι πάρα πολύ άστοχο. Και όλα οι πολιτικές ομάδες προβληματίζουν ε, με αυτό το οποίο τώρα πάμε να αποφασίσουμε. Νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά τι πάμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως με τις ιστορικές και γεωπολιτικές αναλύσεις των περισσότερων συναδέλφων που μίλησαν πριν από μένα. Θα ήθελα κυρίως να αναφερθώ σε ένα θέμα, το πρόβλημα της οικονομικής βιωσιμότητας ε, και σε αυτήν την ένταξη της Μολδαβίας σε μια, ε, σε μια συμφωνία σύνδεσης και ελεύθερου εμπορίου. Ε, πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνουμε ε, για μια οικονομία η οποία υποφέρει τα πάνδυνα κυρίως και μετά το ρωσικό εμπάργο. Αναρωτιέμαι εάν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να δώσουμε μια τέτοια στήριξη στη χώρα αυτή ή μήπως αντιθέτως κινδυνεύουμε να επιδεινωθεί ακόμα ακόμα περισσότερο η πολιτική και η οικονομική κοινωνική κατάσταση στη χώρα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της υπερνηστερίας, συμμερίζομαι απολύτως τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν όσον αφορά το θέμα των διαβατηρίων. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο ε, λαθρεμπόριο ε, όπλων. Ξέρουμε ότι ήταν η βάση της 14ης στρατιάς και ότι από εκεί ξεκίνησε ε, το μεγάλο εμπόριο των όπλων και των βλημάτων κλπ. της ε, ε, ρωσικής ε, στρατιάς. Και είδαμε επίσης ότι έχουν εξαφανιστεί και πύραυλοι με ραδιενεργά ισότοπα στη μύτη τους ας πούμε. Και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια ειδική αντιμετώπιση. Τα θέματα 13, 14 και 15 είναι ιδιαίτερος σημαντικά ε, και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, με μεγάλη προσοχή και από τις δύο πλευρές επίσης είναι σημαντικό να στείλουμε ε, και μια αντιπροσωπεία παρατήρησης και από τη δική μας πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από αυτή του ΟΑΣΕ γιατί πρέπει να έχουμε και εμείς από πρώτο χέρι πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια κι εγώ και ως πρόεδρος αλλά και ως μέλος της Επιτροπής αυτής. Αυτό με τη διαφθορά και τα διαβατήρια ενδιαφέρον μου φαίνεται. Σε ορισμένες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Μάλτα και αλλού μπορεί κανείς με πολλά λεφτά να κάνει επενδύσεις και του δίνουν και διαβατήριο. Αυτό είναι λοιπόν κρατική διαφθορά οργανωμένη, συστηματική και θεσμική. Και αυτό ισχύει μόνο για τους πλουσίους που κάνουν μεγάλες επενδύσεις και αγοράζουν και το διαβατήριο. Αυτό καμιά φορά ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα για να δούμε τι σημαίνει και η ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς κανείς μπορεί να την αγοράσει άμα έχει λεφτά. Λοιπόν, επί της ουσίας, νομίζω αυτό με το άρθρο 49 θα πρέπει να παραμείνει. Είναι μια πάγια διατύπωση, είναι μια φόρμουλα ε, που είναι ένας συμβιβασμός λογικός και έχει να κάνει και με την κατάσταση του δικαίου. Σύμφωνα με το 49, κάθε ευρωπαϊκή χώρα δικαιούται να υποβάλει αίτηση ένταξης. Το εάν θα εγκριθεί αυτή ή όχι, ε, εξαρτάται από τις ε, εκάστοτε συνθήκες που ισχύουν και στη χώρα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορεί να δεχτεί νέα μέλη, αν πληρούνται τα κριτήρια, δεν σημαίνει τίποτα αυτόματο. Είναι μια πάγια ε, διατύπωση που χρησιμοποίησαμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό που έχει να κάνει με τα ιστορικά ζητήματα. Το ανέφερε και ο συνάδελφος Εγκλέσιας. Με όλα αυτά τα πράγματα και τα ιστορικά, ως Γερμανός έχω πάντα κάποιο πρόβλημα. Θυμάστε, η Βεσαραβία ήταν το μέρος όπου έγινε το σύμφωνο Χίτλερ και Στάλιν. Ε, τώρα δεν θα πρέπει να ξυπνήσουμε νέες ε, επιβουλές και ορέξεις της Ρωσίας για τη Δυτική Ουκρανία κτλ. 23 Αυγούστου του 39. Στη βεσαραβία αναφέρεται αυτό. Και ότι δίνεται αυτόματα στην σοβιετική σφαίρα επιρροής. Λοιπόν, αυτά για τα ιστορικά. Και ε, ήταν αυτή η συνθήκη με την οποία οδηγηθήκαμε στον πρώτο, διορθώνει ο Πρόεδρος, στο δεύτερο φυσικά παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε, έχουμε ευθύνη και καθήκον απέναντι στους Μολδαβούς να τους βελτιώσουμε τη ζωή και αυτή η συμφωνία τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη ζωή οι άνθρωποι. Το είπε και ο κύριος Φίλε την περασμένη εβδομάδα, το κατέστησε σαφές για την Ουκρανία. Το 1989 το ΑΕΠ κατά κεφαλήν στην Πολωνία και την Ουκρανία ήταν περίπου παρόμοιο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο οδήγησε σε τετραπλασιασμό σήμερα στην Πολωνία. Και θέλουν και οι Ουκρανοί και οι Μολδαβοί να πάνε εκεί που είναι σήμερα οι Πολωνοί οικονομικά. Και νομίζω είναι και θεμητό αυτό να το ζητούν, να δημιουργηθούν βέβαια οι προϋποθέσεις. Και στο μεταξύ και μόνο φέτος οι εξαγωγές από την Ουκρανία παρά τη δινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν λόγω του πολέμου που τους έφερε η Ρωσία, 15% έχουν αυξηθεί και μόνο φέτος οι ουκρανικές εξαγωγές προς την Ένωση. Αυτά είναι θετικά σημεία και θα πρέπει να το κάνουμε και για τη Μολδαβία αυτό. Υπάρχει οικονομική πρόοδος, υπάρχει και κοινωνική πρόοδος που ανοίγεται με αυτή τη δυνατότητα. Και να μην πάμε στο παλιό σύστημα. Και βέβαια είναι σαφές ότι αυτές οι συμφωνίες και οι συνθήκες βρίσκουν ασύμετρη εφαρμογή. Τι εννοώ, σταδιακά και βαθμιαία υπάρχουν κάποιες προποθέσεις που υποχρεώνεται η Ουκρανία να τις υλοποιήσει ε, όσο μπορεί. Το έχουμε πει αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Εμείς καταργήσαμε τους δασμούς μας για τα ουκρανικά προϊόντα, αλλά το αντίστροφο δεν έχει ισχύσει ακόμα. Και υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για να μπορούν να προσαρμόζονται αυτές οι χώρες στην Τελωνιακή Ένωση και Σύνδεση. Στην συμφωνία μάλλον αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή την τελωνιακή νομοθεσία και το μετασχηματισμό της κοινωνίας, γιατί μόνο έτσι θα φτάσουν εκεί που είναι οι Πολωνοί. Όποιος δεν εξυγχρονίζει την οικονομία ή δεν το επιτρέπεται λόγω ρωσικών ε, επιθυμιών, ε, τότε δεν θα υπάρξει ούτε η κοινωνική πρόοδος, ούτε η οικονομική του κόσμου. Αυτή η λογική νομίζω αποδεικνύεται και κύριε Σόλτς από, στη διαλεκτική πάντα μαθαίνω από εσά. Και πρώτα εξηγείτε ότι το άρθρο 49 ε, δεν θα πρέπει να μπει και μετά εξηγείτε γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί έχει εντηρήσει και επιφυλάξει και η Ρωσία. Δηλαδή, εάν η Μολδαβία δεν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν αρέσει αυτό στη Ρωσία ή γιατί δεν φτάνουν τα εμπορεύματα. Αυτό, όπως γνωρίζουν όλοι οι δίκοι, είναι υποκρισία. Στην Ουκρανία υπήρξε μία τέτοια ε, ρύθμιση αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Ρωσία ποιος έχει ανοιχτά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συμφωνίες. Σήμερα αυτό συμβαίνει ε, και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία συνάδουν απολύτως με τον ΠΟΕ. Να δούμε όμως τι κάνει η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία και πώς ασκεί πίεση σταματάνε τις εισαγωγές. Όλα αυτά είναι απολύτως παράνομα. Τα εμπορικά και οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Ρωσία είναι όλα παράνομα. Και κανείς δεν το αναφέρει αυτό. Και ξαφνικά, τελικά, έρχονται και μας λένε ότι δεν μπορούμε να ε, υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί συνεπείς για να προχωρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε τελική ανάλυση, οι χώρες αυτές αποφασίζουν μόνες τους και η Μολδαβία έχει κυρώσει τη συμφωνία. Με σαφίστατη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και εφόσον έχουν εκείνη κυρώσει, εμείς τι να περιμένουμε. Η δική τους απόφαση είναι κυρίαρχη. Και δεν είναι καθόλου άρον-άρον η διαδικασία. Από το 2007 έχουν γίνει διαπραγματεύσεις και από το 7 μέχρι το 9 δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση, ήταν η προηγούμενη. Που δεν απατώμε, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Πρωθυπουργό κιόλα τότε. Αυτοί κάνανε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Μολδαβίας. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μην ξεχνάμε και το ιστορικό πλαίσιο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά. Λοιπόν, τώρα θα ορίσουμε την προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών ε, ε, αντίστοιχα και παρακαλώ τους συναδελφούς γρήγορα να κάνουν τις τροπολογίες τους πότε είναι 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στις 16 Οκτωβρίου 16 Οκτωβρίου εδώ στην Επιτροπή για να τηρούμε και το χρονικό πλαίσιο. Συμφωνείτε? Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο παρθμόν 6. Παρακαλώ. Δεν σας άκουσα. Ο κύριος Γκάλε. Εγώ ρώτησα Γεωργία πότε θα έρθει. Θα τα πούμε στο διευρυμένο προεδρείο αυτά. Όχι εδώ. Ναι, για να προχωράμε και να προωθούμε τα θέματα. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουμε ένα χρονοδιαγράμμα. 6 Οκτωβρίου για τη Γεωργία η πρώτη συζήτηση, δεύτερη συζήτηση 4 Νοεμβρίου, ψηφοφορία 17 Νοέμβρη και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Μέχρι τώρα έτσι έχει το πλαίσιο κάπως. Αλλά επειδή έχουν στη Μολδαβία εκλογέ, θέλαμε κάπω να επιταχύνουμε τα πράγματα για τη Μολδαβία. Αυτά που σα είπα τώρα ήταν για τη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και κλεισμένο των θυρών. Και παρακαλώ. Τους δημο...